Good afternoon, everybody. Καλησπέρα σε όλους. Έχει πάει τρεις και τέταρτο. Θέλω λοιπόν πως πρέπει να αρχίσουμε. Είναι μια πολύ ευχάριστη στιγμή για μένα. Είμαι στη θέση να καλωσορίσω την Έμιλη στην Επιτροπή Αναφορών, η οποία θα μας παρουσιάσει το όραμά της σε αυτήν την ακρόαση. Σκοπός τη ακρόαση αυτή είναι να έχουν οι ευρωβουλευτέ τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την καταλληλότητα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο έχει έναν, μία μόνο υποψήφια για τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Όπως ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο πρόεδρο Σούλτ, είναι η Έμιλι Οράιλι, είναι λοιπόν αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναφορών να δημιουργήσει μία πλατφόρμα όπου τα ενδιαφερόμενα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα θέσουν ερωτήσεις στις οποίες η υποψήφια θα απαντήσει. Η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε, βασισμένη στις συστάσεις της Επιτροπής μας, ότι η εκλογή θα γίνει το μεσημέρι της Τρίτης στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, δηλαδή στις 16 του μήνα. Μετά από τη σημερινή ακρόαση, η δήλωση της κυρίας O'Reilly θα δημοσιευθεί σε όλες τις γλώσσες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Διαμεσολαβήτριας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ερωτήσεις θα ακολουθήσουν την μέθοδο DEONT και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε εκπροσώπους από όλες τις πολιτικές ομάδες, αν δεν κάνω λάθος σχεδόν από όλες. Θα αρχίσουμε λοιπόν με τις μεγάλες πολιτικές ομάδες, όμως η κυρία Οράλη θα κάνει τώρα τη δήλωσή της και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για, την... για το εγκάρδιο Αγαπητά μέλη, έχω την τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας ως υποψήφια για τον επαναδιορισμό μου στο αξίωμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Θα ήθελα να αναφερθώ στο το έργο μου κατά το πρώτο έτος της θητείας μου και να σας παρουσιάσω το όραμα και τη στρατηγική μου για το θεσμό για την ερχόμενη πενταετία. Αυτή είναι η έβδομη φορά που σας απευθύνω ομιλία ως διαμεσολαβήτρια. Με Κάθε φορά έχω αποκομίσει ωφέλη από την εμπειρογνωμοσύνη σας, τις συμβουλές και τη στήριξή σας, καθώς και από το προσωπικό που στηρίζει το έργο σας. Αυτές οι ακροάσεις των επιτροπών, όπως και οι πολυάριθμες διμερείς συναντήσεις μας, με έχουν βοηθήσει να κατανοήσω καλύτερα το κοινό μας έργο και έχουν συμβάλει άμεσα στη διαμόρφωση της στρατηγικής που έχω αναπτύξει για το θεσμό του διαμεσολαβητή. Η ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών μου και του Κοινοβουλίου θα καθορίσει τον βαθμό επιτυχίας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας της διοίκησης προς όφελος των πολιτών της Ένωσης. Ω τρίτη Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, αρμοδιότητά μου είναι να αναπτύξω περαιτέρω το έργο του διαμεσολαβητή και να διασφαλίσω ότι θα εξακολουθεί να είναι επιτυχημένη. Στην τελετή ορκομοσία πέρυσι στο τμήμα μείζωνο συνθέσεω του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο, δήλωσα ότι οι πολίτε τη Ευρώπη δεν ζητούν πλέον απλώ τα λόγια και τα όμορφα λόγια των συνθήκων και των χαρτών, αλλά την καθημερινή του μεταφορά σε πολιτικέ και δράσει που έχουν αντίκτυπο στην πραγματική του ζωή. Η φιλοδοξία μου είναι απλή. Να βοηθήσω τα θεσμικά όργανα τη Ένωση να δίνουν τον καλύτερό του σε αυτό να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που έχουν και που έχουν οριστεί για αυτά από τις συνθήκες και τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το περασμένο έτος ασχολήθηκα με την μετατροπή των λόγων σε πράξεις και η στρατηγική μου έχει τρεις στόχους. Εξασφάλιση της συνάφειας, αύξηση της προβολής και επίτευξη μεγαλύτερου αντικτύπου. Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε περαιτέρω στη διάρκεια του έτους, μετά από πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις και σε εσωτερικό και σε εξωτερικό επίπεδο. Πρόσφατα δημοσίευσα την πενταετή στρατηγική μας με τίτλο «Προς το 2019», την οποία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας. Αρχικά, για να ξεκινήσω την εκτέλεση της στρατηγικής, ξεκίνησα έναν εσωτερικό έλεγχο των ε, διαδικασιών και πρακτικών των υπηρεσιών του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Αυτό οδήγησε σε πολλέ εσωτερικέ αλλαγέ, όπω για παράδειγμα την εισαγωγή ενό σύγχρονου συστήματο διεκπαιρέωση καταγγελιών. Είναι μια διεργασία που ξεκίνησε προκάτοχό μου και θα μα επιτρέψει να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη διεκπαιρέωση. Στις αλλαγές αυτές επίσης συγκαταλέγεται η επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο συντάσσουμε τις αποφάσεις μας, η επανεξέταση των κύριων δικτών επιδόσεων και των διεργασιών έρευνας και καταγγελίας, τα οποία θα μας επιτρέψουν να εντοπίζουμε έγκαιρα τις σημαντικές υποθέσεις. Πιστεύω πως αυτές οι αλλαγές θα βελτιώσουν συνολικά τις υπηρεσίες μας προς τους πολίτες. Οι υπηρεσίε μα διαθέτουν λιγότερου από 100 υπαλλήλου. Θεωρώ λοιπόν καθήκον μου να χρησιμοποιήσω με το βέλτιστο δυνατό τρόπο του διαθέσιμου πόρου. Και για να είμαστε όσο το δυνατόν κοντύτερα στις, ε, στους πολίτες μας, αξιοποίησα περισσότερο την εξουσία να κοινώ έρευνε δημοσίου συμφέροντος χωρίς αυτές να βασίζονται απαραίτητα σε συγκεκριμένη καταγγελία. Για το σκοπό αυτό διόρισα μια συντονίστρια αυτεπάγγελτων ερευνών, η οποία έχει ως αρμοδιότητα να συντονίζει μαζί με τους συναδέλφους της τις αυτεπάγγελτες έρευνες και να εξασφαλίζει την ταχεία και πατάλληλος μετακή διεκπαιρέωσή τους. Το έτος αυτό ξεκινήσαμε αυταπάγγελτες έρευνες για τη διαφάνεια των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων για την Συμφωνία TTIP, τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα εφαρμόζουν τους νέους κανόνες σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χειρίζεται την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, τα ε, προγράμματα του Ταμείου Συνοχής και με τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η τήρηση του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την Frontex. Δύο ακόμα σημαντικές έρευνες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χειρίζεται συγκρούσεις συμφερόντων όταν οι υπάλληλοι της αποχωρούν για να εργαστούν αλλού και τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων στηρίζει τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για την διαφάνεια όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές. Για να επιτύχουμε μεγαλύτερη προβολή, εστίασα τις προσπάθειές μου στη βελτίωση της προβολής του έργου σε εσά, του ε, εκλεγμένους, τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό. Σχολιαστές και αναλυτές των μέσων ενημέρωσης βεβαιώνουν ότι η στρατηγική έχει σημαντικό αντίκτυπο, καθώς και λεπτομέρειες των υποθέσεών μας εμφανίζονται πλέον τακτικά στα μέσα ενημέρωσης των Βρυξελών αλλά και των κρατών μελών και σε άλλα μέρη. Παράλληλα πλέον λαμβάνετε και εσεί σύνοψη του έργου μα και ελπίζω ότι έχω αποδείξει την προθυμία μου για συνεχή ε, διάλογο μαζί σας για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Δώσαμε επίση έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τριπλασιάσαμε τους ε, οπαδούς μας στο Twitter σε διάστημα ενό έτου. Πολλοί από εσά έχετε δει τη νέα μορφή τη ετήσια έκθεσή μα, η οποία έχει κατατεθεί στο Κοινοβούλιο. Η επικοινωνιακή μου στρατηγική βασίζεται στην πεποίθηση ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούμε το έργο μας ως το δυνατόν περισσότερο και με μεγαλύτερη προσβασιμότητα για να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να προσφεύγουν σε εμά όταν παρατηρούν περιστατικά εικαζόμενης κακοδίκησης τα οποία θεωρούν ότι χρήζουν διερεύνησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα επικοινωνίας η οποία αγκάλιασε τη νέα στρατηγική με μεγάλο ενθουσιασμό, ενέργεια και δημιουργικότητα. Πολλέ από τι νέε μα έρευνε βρίσκονται εν εξέλιξη. Πιστεύω ότι η νέα στρατηγική έχει ήδη αποτελέσματα και είμαι ευγνώμων σε όλου με του οποίου συνεργάστηκα για τη θετική συμμετοχή του. Το περασμένο Δεκέμβριο λάβαμε τη θετική ανταπόκριση τη Επιτροπή για δύο σημαντικέ υποθέσει. Η μία αφορούσε αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε σχέση με κρατικέ ενισχύσει σε συγκεκριμένου συλλόγου επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ενώ η δεύτερη αφορούσε η καζόμενη σύγκρουση του πρώην Προέδρου της ΑΝΤΟΚ Επιτροπής Δεοντολογίας για Επιτρόπους. Ο Πρόεδρος παρετήθηκε μετά την παρέμβασή μου και η Επιτροπή έκτοτε προσέδωσε μεγαλύτερη διαφάνεια ε, στο έργο της ΑΝΤΟΚ Επιτροπής Δεοντολογίας. Νομίζω ότι η παρέμβαση των υπηρεσιών μας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων με συμμετοχή ενδιαφερομένων βουλευτών και της κοινωνίας των πολιτών συνέβαλε στο να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει παναχώρηση από τη νέα πολιτική διαφάνειας όπως φάνηκε να συμβαίνει νωρίτερα φέτος. Επιπλέον, μετά από κοινή παρέμβαση ενδιαφερομένων Ευρωβουλευτών και της κοινωνίας ε, των ε, πολιτών και μετά από έρευνες των υπηρεσιών μας όσον αφορά την έλλειψη διαφάνεια σε σχέση με την διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου για τις ε, συνεμιλίες με την TTIP, το Συμβούλιο δημοσιοποίησε την εντολή για ευρύτερο δημόσιο έλεγχο. Τέλος, μετά τη συνεδρίαση με τον πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Ντράγκη, νωρίτερα φέτος η ΕΚΤ ζήτησε τη Συμβουλή των Υπηρεσιών μας σχετικά με τη νέα πολιτική δεοντολογίας και εκφράζω την την ικανοποίησή μου. Όπως ε, είχα πρόεδρο ε, με τον κύριο Μάριο Ντράγκη νωρίτερα ε, και τώρα μου ζητήθηκε να τον συμβουλεύσω για τη νέα αυτή πολιτική διοντολογία και χαίρομαι για το θέμα αυτό. Όπως ξέρετε, η ΕΚ διαθέτει νέες εξουσίες τραπεζικής εποπτείας και για τον λόγο αυτό αύξησε σημαντικά τον αριθμό των υπαλλήλων της. Θα πρέπει λοιπόν ε, να έχει υψηλό επίπεδο δεοντολογίας. Έχω την τιμή να εκλεγώ και πάλι, εάν έχω την τιμή να εκλεγώ και πάλι από το Κοινοβούλιο, θα ήθελα να συνεχίσω την ανάπτυξη αυτής ε, της στρατηγικής στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Η δύναμη του διαμεσολαβητή στην άσκηση δημοκρατικής εποπτείας της δίκησης εξ ονόματος των πολιτών είναι ισχυρή μόνο στο βαθμό που είναι ισχυρός και ο δεσμός του με τον Κοινοβούλιο. Τις τελευταίες εβδομάδες άκουσα προσεκτικά τι απόψει τη νέα Επιτροπή και ιδίω εκείνων που θα ηγούνται αυτού του σημαντικού θεσμικού οργάνου στα επόμενα δύσκολα έτη. Οι δεσμεύσει για μεγαλύτερη διαφάνεια, ανοιχτό χαρακτήρα, λογοδοσία και εμπιστοσύνη μου φάνηκαν ενθαρρυντικέ και δεσμεύομαι να συνεργαστώ στο δυνατόν πιο στενά με την Επιτροπή για να τη βοηθήσω στην επίτευξη των στόχων αυτών. Ολοκληρώνοντα, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω και πάλι πόσο είμαι εντυπωσιασμένη από τα υψηλά πρότυπα Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση των χιλιάδων αφοσιωμένων ατόμων που εργάζονται στα θεσμικά όργανα. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών εργάζονται εργάζονται σκληρά για να επιτύχουν υψηλά πρότυπα στην εργασία τους και διαπνέονται από πραγματική δεοντολογία δημόσιας δίκης. Εν τούτης, όπως γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η εμπιστοσύνη στην διακυβέρνηση δεν είναι ε, σημαντική. Οι λαοί της Ευρώπης θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στους ειδίκης όταν αρχίσουν να βλέπουν θετικές αλλαγές που απορρέουν από τις αποφάσεις αλλαγές για τις οικογένειές τους στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, αντίθετα με τα περισσότερα εθνικά κράτη στην Ευρώπη, τα οποία έχουν νομιμοποιήσει στα μάτια των πολιτών τους, η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμα επιτύχει το υψηλό επίπεδο νομιμοποίησης που θα έπρεπε στα μάτια πολλών Ευρωπαίων. Γι' αυτό θα πρέπει η διοίκηση να έχει όχι μόνο την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, αλλά και τα υψηλότερα πρότυπα διοντολογίας, διαφάνειας, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας. Η αποστολή μου Διαμεσολαβήτρια είναι να συνεργαστώ τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς για να βοηθήσω στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αν εσείς οι ευρωβουλευτές με εμπιστευτείτε με την ψήφο σας για να συνεχίσω το έργο μου, υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να φέρω σφαίρα στην αποστολή μου και θα διευθύνω το έργο των υπηρεσιών μου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τηρώ τη δέσμευσή μου προς εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε σε όλα τα θέματα. Απαιτείται να αντιμετωπίσουμε με ευρωπαϊκό τρόπο τα προβλήματα των πολιτών ανεξαρτήτως του οργάνου το οποίο εκπροσωπούμε. Και είναι θετικό το ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας. Ερωτήσεις. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Βαλένζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Οράιλη. Δεν είναι πολλά τα παρόντα μέλη. Αυτό δεν είναι ένδειξη ασέβειας, αλλά οργανώθηκε για να αποδείξετε τις ικανότητές σας και σε ό,τι με αφορά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το κάνετε. Έχω όμως έξι ερωτήσεις. Παρακαλώ αν μπορείτε να απαντήσετε. Η πρώτη ερώτηση. Η βασική ανησυχία, ή μάλλον ποια είναι η βασική ανησυχία των πολιτών και τι μπορεί να γίνει για να μικρύνει η απόσταση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά όργανα και τους πολίτες πώς μπορείτε να βελτιώσετε την καλύτερη κατανόηση του τι κάνει και του πώς δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη ερώτηση, ο Ομπουτσμαν έχει μηχανισμούς στην διάθεσή του και μέσα έτσι ώστε να περνάει και να ακούγεται το μήνυμά του. Ποιοι είναι οι στόχοι σας σε σχέση με την πολιτική σας στήριξη από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της δεύτερης περίοδου σας. Τώρα και στην δική μου έκθεση και γύρω από την έκθεση πολλά μέλη ασχολήθηκαν με το θέμα της έλλειψης συμμόρφωσης. Γνωρίζω ότι η έκθεση για τη συμμόρφωση είναι υποπροετοιμασία. Μπορείτε παρακαλώ να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχει παράλληλα και το επόμενο θέμα για το TTIP να σας συγχαρώ γι' αυτό γιατί ξέρω ότι και χάρη στη δική σας παρέμβαση εδώ και μία εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δημοσιεύσει περισσότερα κείμενα υποδιαπραγμάτευση και να ανοίξει την πρόσβαση σε άλλα έγγραφα. Ξέρω ότι εσείς έχετε πάρει πολλές απαντήσεις για τις δημόσιες διαβουλεύσεις για τα TTIP. Ε, μπορείτε να μας πείτε σε ποια φάση βρίσκονται οι διαβουλεύσεις. Επόμενη ερώτηση σχετικά με την Τρόικα. Ποια είναι η άποψή σας για τις δραστηριότητες γύρω από την Τρόικα. Υπάρχουν ορισμένα μέλη στην Επιτροπή μας που ενδιαφέρονται ιδιαίτερως. Θεωρείτε ότι το θέμα της Τρόικα θα πρέπει να ερευνηθεί ο ρόλος της Επιτροπής, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και τέλος, είναι κάτι στο οποίο αναφερθήκατε βέβαια, το θέμα της αναπηρίας. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των αναπήρων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που έχετε θέσει σαν στόχο. Να σας συγχαρώ για την αυξημένη παρουσία σας επίσης και στα κοινωνικά μέσα. Πώς θα ισορροπήσετε ανάμεσα στο παραδοσιακό κανάλι επικοινωνίας και στα νέα κανάλια επικοινωνίας, γιατί υπάρχουν ε, κάποιες ανησυχίες για τον αποκλεισμό αυτών οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα νέα μέσα. Πρέπει να υπάρξει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στα παλιά και τα νέα μέσα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ κύριε Βαλένσο για τις ερωτήσεις σας. Είναι ακριβώς ο πυρήνας αυτών που κάνω για την επικοινωνία και τη γεφύρωση της διαφοράς ανάμεσα την απόσταση ανάμεσα στην Ένωση και τους πολίτες της. Είναι μια δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουν όλα τα όργανα. Ενθυμούμε πριν μερικούς μήνες και ήμουνα έξι μήνες ομπουτσμαν ε, τότε και πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπω το πόσο ε, εμπλέκεται κανείς και να πηγαίνω μετά στο σπίτι μου και να βλέπω ότι η απόσταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι είναι κάτι που σε κάνει να σκέφτεσαι πραγματικά πώς είναι τα πράγματα. Ήταν περίεργη η αίσθηση γιατί ταυτόχρονα τα τρία μέλη της Τρόικα ήταν σε ένα ξενοδοχείο στο Δουβλίνο και ε, πήγαιναν κάθε μέρα ε, στα κτίρια της κυβέρνησης να μας λένε το τι έπρεπε να κάνουμε. Ε, γι' αυτό δείχνει ότι η γέφυρα δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη και είναι λογικό να διαρωτώνται οι πολίτες γιατί συνέβη κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό λοιπόν. Υπάρχει και θέμα γλώσσας, θέμα μεταφράσεων, θέμα συμβιβασμών που οδηγεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις Πραγματικά πάρα πολλές φορές ε, ε, ε, η ουσία των νομοθετικών ρυθμίσεων δεν γίνεται αμέσως αντιληπτή και αυτό είναι ένα θέμα. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε τη συνείδησή μας για να δούμε το τι πράγματι κάνουμε. Τώρα το τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Τώρα νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο αυτή τη στιγμή περνά έχει σχέση με τη μεγαλύτερη ανάγκη εμπλοκής των πολιτών, ιδιαίτερα στον τομέα της διαφάνειας. Νομίζω ότι αυτή είναι μια έννοια στην οποία πρέπει να σταθούμε. Και ήδη από χθε έχουμε λεπτομέρειες των συναντήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι επίτροποι σε σχέση με συμφέροντα επιχειρηματικά κτλ. Έχουμε επίσης προτάσεις που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα για μεγαλύτερη διαφάνεια και στην ουσία οι διαπραγματεύσεις για το TTIP είναι η ένδειξη η οποία θα μας δώσει να καταλάβουμε αν πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περάσει σε μια νέα λειτουργία. Φυσικά και οι κυβερνήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξουν για τον τρόπο με τον οποίο ενημερώνουν και μέσα στα κοινοβούλια, έχουν ειδικέ επιτροπές. Ε, νομίζω ότι εγώ από τη δική μου πλευρά η μεταφορά του μηνύματός μου προς τους πολίτες μέσω του κοινοβουλίου, των κοινοβουλίων, είναι ο στόχος, είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια παροιμία στη γλώσσα μου που λέει ότι αν πέσει ένα δέντρο μέσα στο δάσος και δεν το έχει δει κανείς, έπεσε τελικά αυτό το δέντρο. Λοιπόν, το θέμα είναι να φαίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Τώρα για την πολιτική στήριξη, την πολιτική εξουσία, εγώ δεν έχω πολιτική εξουσία αυτής. Ξέρετε ότι εγώ από αυτά τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια της επιλογής μου ότι εκτιμώ ιδιαίτερο τις εργασίες σας και εγώ μίλησα πέρυσι αναλυτικά για την ανάγκη συνάντησης με τις επιμέρους κοινοβουλευτικές επιτροπές και τα μέλη του Κοινοβουλίου όταν ήμουνα εθνική ομπουτσμαν. Εθνική Διαμεσολαβήτρια, ήδη παρακολουθούσα τις εργασίες σας και έβλεπα τις διαφορές που υπάρχουν ε, ανάμεσα στη χώρα μου και ανάμεσα σε αυτά τα οποία συνέβαιναν εδώ. Και επέμεινα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη με τη δική σας επιτροπή ε, στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, το θέμα της μη συμμόρφωσης είναι κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εγώ έχω πει ότι δεν είμαι ικανοποιημένη από το ποσοστό συμμόρφωσης, το οποίο είναι γύρω στο 80% στην παρούσα φάση. Φαίνεται πολύ ψηλό, αλλά σε ορισμένες χώρες ο αριθμός είναι ανάμεσα σε 90 με 100% και είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα εγώ να αλλάξω την λειτουργία της δικής μου υπηρεσίας. Ε, μερικές φορές ε, το να τοποθετείτε στο αρχείο ε, ένα αίτημα, μια αναφορά, δεν σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πολλές φορές είναι η αρχή της διαδικασίας και γι' αυτό τους επόμενους έξι μήνες και τον επόμενο χρόνο εφόσον επανεκλεγώ θα προσπαθήσω να δω ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους θέλω να δω να εκπληρούνται. Και θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα ιστορικό των κινήσεών μου μέχρι τώρα για να διασφαλίσω τη μέγιστη δυνατή συνόρφωση. Θα πρέπει επίσης ε, να δουλέψουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πιο συνεργατικό τρόπο. Ε, το να στείλω μια επιστολή και να μου απαντήσουν και τα λοιπά ε, δεν είναι κάτι το επαρκές. Νομίζω ότι το προσωπικό μου σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι ερευνούν, θα πρέπει να συνεργάζονται και να εργάζονται με τους ομολόγους τους στις διάφορες εξωτερικές υπηρεσίες και στην Επιτροπή για να καταλαβαίνουν τι περί τίνος πρόκειται και για να δείξουμε ότι από κοινού μπορούμε να διασφαλίσουμε μια σωστή κατάληξη για τον πολίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να δω να αυξάνεται λοιπόν η συμμόρφωση για το TTIP. Έχουμε 300 γραπτές απαντήσεις, έχουμε και 6.000 mail γύρω από αυτά θα ήθελα να μπορέσω να στείλω κάποιες συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να γίνει η εργασία της ΠΟΔ διαφανής. Ε, πάντα βέβαια ένα τμήμα των διαπραγματεύσεων πρέπει να παραμένουν σε ιδιωτικό επίπεδο τουλάχιστον για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ε, πρέπει τα στοιχεία αυτά να παραμένουν περιορισμένα έτσι ώστε να μπορεί να προχωράει η διαπραγμάτευση μερικές φορές. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αντιμετωπίζει πλέον το θέμα βλέπει ότι έχει μεγάλη σημασία και οι προτάσεις τις οποίες έκαναν τις τελευταίες μέρες αυτό αποδεικτείων. Υπήρξε μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα το πρωί σε σχέση με τις προτάσεις τις οποίες τους έχω κάνει. Θα τις μελετήσω, είπαν ότι θέλουν να εργαστούν μαζί μου εγώ θα κάνω τις τελικές μου προτάσεις τον Ιανουάριο. Τώρα για την Τρόικα. Υπάρχουν επανειλημμένα αφορμές που έχω μιλήσει σε εσά και σε άλλες επιτροπές και ατομικά σε βουλευτές ήδη και την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με την Τρόικα. Προέρχομαι από μια χώρα η οποία βίωσε τις επιπτώσεις. Η Ιρλανδία δεν έχει υποφέρει με τον ίδιο τρόπο άλλες χώρες ε, που έχουν βιώσει άλλες χώρες, η οικονομική περιθωριοποίηση ήταν αποτέλεσμα των πολιτικών μερικές φορές που επέβαλαν οι κυβερνήσεις επειδή το επέβαλε η Τρόικα. Αυτό δεν το βιώσαμε στο ίδιο επίπεδο με άλλες χώρες. Θα ήταν λάθος όμως να υποσχεθώ ότι θα κάνω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω εγώ θα πρέπει να εργαστώ στα πλαίσια των ορίων μου και της εμβέλειάς μου. Η Τρόικα είναι ένα υπερεθνικό σώμα. Ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι βέβαια κοινοτική, η Επιτροπή είναι κοινοτική, αλλά το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ δεν είναι κοινοτικό όργανο. Και γενικότερα υπάρχει αίσθηση ότι στην Ιρλανδική περίπτωση η οικονομία βέβαια ανακάμπτει στην παρούσα φάση, ενώ άλλες χώρες δεν ήσαν τόσο τυχερές. Πάντως αισθάνομαι και από αυτά που λέει το Κοινοβούλιο και από πολίτες της χώρας μου ότι υπήρξε μια αίσθηση του «Μα ποιοι είναι αυτοί οι τύποι, σε ποιον είναι υπόλογοι» και τίθεται ένα θέμα εδώ ευθύνης, αναφοράς ευθύνης, έτσι ώστε ο κόσμος να καταλάβει ε, ακριβώς πώς λειτουργεί το σύστημα. Συζητούσα με έναν Ευρωβουλευτή την προηγούμενη εβδομάδα και είπα ότι αν υπάρχει πράγματα ένας τομέας της εργασίας της Τρόικα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κακοδιαχείριση και κακή διοίκηση εις βάρος των ευρωπαϊκών οργάνων, εγώ μπορώ να ασχοληθώ με αυτό και το θέμα της διαφάνειας είναι ένα θέμα βέβαια. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι υπάρχει ένα θέμα, στο πλαίσιο αυτό έτσι ώστε η υπηρεσία μου στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχει και των αρμοδιοτήτων της να μπορέσει να ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά θα ήταν λάθος και ανάρμοστο για μένα να υποσχεθώ πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κάνω και που δεν είναι δική μου δουλειά. Τώρα, εγώ είμαι παραδοσιακή δημοσιογράφος, εγώ ξεκίνησα με με γραφομηχανές, ούτε τηλέφωνα κινητά είχα, ούτε τίποτα. Αντέγραφα την, το, το κείμενό μου με καρμπών. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία να συνδυάζουμε τις μορφές επικοινωνίας. Φυσικά και τα νέα μέσα είναι απαραίτητα, είναι η πραγματικότητα σήμερα, είτε σας αρέσει είτε όχι φιλοσοφία μου είναι ότι θα πρέπει να είμαστε όσο πιο δεκτικοί μπορούμε, όσο πιο προσβάσιμοι μπορούμε και να επικοινωνούμε με τρόπους οι οποίοι θα καταστήσουν όλους μας ικανούς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν όσοι έχουν παράπονα μπορούν να μας στείλουν mail, μπορεί να μας γράψουν, μπορεί να μας τηλεφωνήσουν. Με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε προσβάσιμοι και αν έλθουν σε μένα μέλη του Κοινοβουλίου ή κάποιοι πολίτες που έχουν δυσκολία επικοινωνίας μαζί μας ή κάποιοι συμπολίτες τους έχουν δυσκολία επικοινωνίας, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην Σολεδάδ Ρούις, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Να ξεκινήσω συγχαίροντας λοιπόν την Ombudsman και την μελλοντική προφανώς, όχι μόνο την παρούσα, γιατί νομίζω ότι η υποψηφιότητά σας είναι δείγμα ακριβώς της πολύ καλή δουλειάς που κάνατε στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα κάποιες διαφημίσεις να κάνω και να θέσω μια ερώτηση. Θα θέλω να χαιρετήσω την ικανότητα ε, αντιμετώπισης ε, ενός θέματος πολύ πάρα πολύ σημαντικά θέματα ε, με τα οποία ασχολούμεθα. Θα ήθελα αν προβλέπετε να πάρετε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες με τα ευρωπαϊκά όργανα. Διότι είναι σαφές ότι και μετά από αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος κ. Βαλέσα είναι σημαντικό να είναι σωστά ενημερωμένος ο πολίτης ιδιαίτερα στα πλαίσια της κρίσης. Έχει σημασία λοιπόν να προσπαθήσουμε να είμαστε σε επαφή σαν ευρωπαϊκά όργανα με τους Ευρωπαίους πολίτες. το τι ακριβώς γίνεται με τις φαρμακευτικές ουσίες και με τα φάρμακα. Δεν ξέρω αν εδώ τίθεται ένα θέμα δικαιώματος των πολιτών, αλλά το θέμα είναι να δούμε τι συμβαίνει με την βιωσιμότητα των συνδικάτων ε, των συστημάτων ε, πρόνοιας ε, ιδιαίτερα με τις πιέσεις που ασκούν οι μεγάλες φαρμακευτικές, βιομηχανικές ή μη μονοπωλιακές επιχειρήσεις στα συστήματα υγείας. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο να πάρετε κάποια μέτρα έτσι ώστε να ερευνήσετε τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία επανειλημμένα τίθενται. Τώρα, και θα ήθελα να χαιρετήσω την προσπάθεια διαφάνειας την οποία έχετε ξεκινήσει, όπως επίσης και την δυνατότητα προσβασιμότητας την οποία επιδεικνύεται και μέσα, το, μέσα από το καινούριο πόρταλ σας και μέσα των επιμέρους δημοσίευσεών σας. Μήπως λοιπόν θα θεωρούσατε απαραίτητο να συνεχίσετε στον δρόμο αυτό ε, έτσι ώστε να, να έρθετε κοντά στις κοινότητες οι οποίες έχουν περισσότερα προβλήματα, είναι οι πιο ευάλωτες, σαν παράδειγμα ε, το θέμα της παιδικής ηλικίας, το θέμα των παιδιών. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ότι τα παιδιά είναι, πέφτουν θύματα πολύ κακής μεταχείρισης και γι' αυτό αναρωτιέμαι αν υπάρχει δυνατότητα ε, να δοθεί ε, στην, ε, μια ειδική θέση στην προσπάθεια που κάνονται για την παιδική ηλικία, για τους νέους και τα παιδιά. Επίσης το θέμα των αναπηριών να είναι μια κατηγορία ανθρώπων η οποία θα πρέπει να μας απασχολήσει έτσι ώστε να μπορούν σαν παράδειγμα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες σας για θέματα πάρα πολύ σημαντικά και μάλιστα υπάρχουν ειδικότερα προβλήματα για αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα κυρίως... Οι ε, προβλήματα διανοητικά όπως επίσης και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτοί οι οποίοι τους φροντίζουν Λοιπόν, ε, το θέμα είναι ότι το σύνολο των ε, αποφάσεών σας και των σχολείων σας ε, να είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι απαραίτητο, όχι μόνο στα αγγλικά, γιατί αλλιώς αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο, ένα πολύ κρίσιμο εμπόδιο, ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα. έτσι δεν μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, ε, μου κάνει εντύπωση ότι η έκθεση την οποία ψηφίσαμε σήμερα το πρωί που είναι μια γυναίκα έχει πάρα πολύ ε, μεγάλη σημασία να μιλήσουμε με μια ενιαία γλώσσα για να μπορέσουμε να σας ονομάζουμε σωστά. Λοιπόν, ε, στα ισπανικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε θα έλεγα μια φράση η οποία μεταφράζεται η προάσπιση των συμφερόντων του λαού ή προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών. Έχει σημασία λοιπόν να προσέξουμε την ορολογία. Τώρα για το θέμα της διαφάνειας και των, της υπηρεσίας σας και των υπολείπων κοινωτικών οργάνων έχει μεγάλη σημασία να το επιδιώξετε στις επαφές σας με την Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη και ίσως θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες εγγυήσει για την απάντηση από πλευράς της Επιτροπής και των κρατών μελών στις ερωτήσεις σας και στα σχόλιά σας έτσι ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο η ανεξαρτησία σας αλλά και η έγκαιρη απάντηση στις αναφορές τις οποίες καταθέτουν οι συμπολίτες μας. ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, κυρία Κράσαν Ρούις. Αναφερθήκατε στην αρχή για το πώς έγινε αντιληπτή η κρίση. Φυσικά και η κρίση έγινε αντιληπτή από διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο και ήταν πολύ πιο έντονη σε ανθρώπους που ήταν ήδη φτωχοί, που είχαν χάσει τις δουλειές τους, που ήταν άτομα με αναπηρία, δηλαδή σε άτομα τα οποία ήταν όντως ε, μειονεκτική θέση ή ήταν περιθωριοποιημένα. Πιστεύω πως ε, έργο του Κοινοβουλίου είναι να καταστήσει πιο ορατή την κατάσταση. Πιστεύω πως Υπήρχε η αίσθηση από τα μέσα της κρίσης έως και τώρα ότι η κρίση ήταν κάτι το καθαρά δημοσιονομικό, αφορούσε καθαρά και μόνο την αγορά και έλειπε το κοινωνικό στοιχείο, έλειπε το πώς ε, είχε, το τι αντίκτυπο είχε η κρίση στους ε, πολίτες και πιστεύω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λαμβάνουν αποφάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το νέο επενδυτικό ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, θα υπαγορεύσουν ε, τρόπον την, την δέσμευσή τους. Θα περιγράψουν τη δέσμευσή τους για την αντιμετώπιση της κρίσης και Θυμάμαι ότι ο Επίτροπος κύριος Τίμερμανς, όταν μίλησε για την πρωτοβουλία των πολιτών, που είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε ακριβώς για να γεφυρώσει αυτό το κενό ανάμεσα στους πολίτες και τα θεσμικά όργανα. Και όπως ξέρετε, Καμία από τις ε, προτάσεις δεν, έγιναν, ε, δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή, ακόμα και προτάσεις που συγκέντρωσαν πολλές υπογραφές. Ο κύριος Τίμερμανς, λοιπόν, είπε ότι θεώρησε πως η πρωτοβουλία των πολιτών έγινε αντιληπτή περισσότερο σαν νομικό μέσο και όχι σαν πολιτικό μέσο και πιστεύω πως πραγματικά θέλησε με τον τρόπο αυτό να μας επιστήσει την προσοχή στον στόχο της πρωτοβουλίας των πολιτών και στο να αναρτηθούμε ποια είναι η θέληση και η πολιτική θέληση και οι δυνατότητες που έχουν τα θεσμικά όργανα, αλλά και η πρακτική οργανωτική θέληση που υπάρχει. Και πιστεύω πως δεν μιλώ πολιτικά όταν λέω ότι η πρωτοβουλία των πολιτών είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Εγώ έχω κάνει κάποιες ε, σαφείς προτάσεις και ελπίζω να συνεισφέρουμε σημαντικά Επίσης, ε, μιλήσατε για το μονοπόλιο των φαρμακευτικών και εδώ υπάρχουν θέματα πολιτικής, πολύ σοβαρά θέματα πολιτικής τα οποία πρέπει να συζητηθούν και η Συμφωνία TTIP ανήκει σε αυτά. Και σίγουρα υπάρχει κάποια δυνατότητα επιρροής μέσω του Μητρώου Διαφάνειας ε, στο οποίο θα καταγράφονται τα λόμπι έτσι ώστε να φαίνεται ποιος επηρεάζει τι και σε τι θέση βρίσκονται οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. Υπάρχουν κάποιες ε, αλλαγές οι οποίες έχουν ανακοινωθεί σχετικά με το Μητρό Διαφάνειας και τα θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κάνει κάποιες δεσμεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα, έχει δεσμευτεί ότι οι ανώτεροι διευθυντές των ε, γενικών διευθύνσεων θα πρέπει να διαθέτουν στη δημοσιότητα έναν κατάλογο με το ποιους ε, συναντούν. Πιστεύω πως έχει έρθει η στιγμή να περάσει το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν πρέπει να δείχνουν δυσπιστία απέναντι στα θεσπικά όργανα. Διότι υπήρχε η τύπωση ότι κρύβονται πράγματα μόνο και μόνο για να μην ε, γίνουν γνωστά. Όμως έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πάρα πολλά έγγραφα, τα οποία δεν οδήγησαν και σε κάποιες συνταρακτικές εξελίξεις. Πιστεύω πάντως, όπως και να έχει, πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δεσμευτεί για ακόμα περισσότερη διαφάνεια, για όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των ε, παιδιών, σε πολλές χώρες και στη δική μου χώρα υπάρχει ειδικό γραφείο του διαμεσολαβήτη για τα παιδιά και το γραφείο αυτό και ο διαμεσολαβητής για τα παιδιά διορίζεται εν μέρει και από την κυβέρνηση μετά από ακρόαση και από τα κοινοβούλια. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ε, δυνατότητα αυτού του δικτύου διαμεσολαβητή για τα παιδιά. Μπορούμε να διοργανώσουμε και κάποιες εκδηλώσεις όπως για παράδειγμα κοινοβούλιο για παιδιά ή παρόμοιες εκδηλώσεις. Πρέπει να δούμε τα δικαιώματα των παιδιών ως άτομα και όχι ως μέρος της οικογένειας. Τώρα, όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, πέρυσι διορίσαμε έναν ε, αρμόδιο για θέματα ανθρώπων με αναπηρία και πιστεύω κιόλας ότι η πρώτη συνθήκη που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα ήταν η συνθήκη για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Πιστεύω πως τα θεσμικά όργανα συμμορφώνονται με τις επιτάξεις για τα άτομα με αναπηρία και ως ε, διαμεσολαβήτρια της Ιρλανδίας είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με τα άτομα αυτά. Ε, μία από τις ε, πρώτες μου ενέργειες ήταν η δημιουργία πρόσβασης στα άτομα με αναπηρία στα κτίρια μας και στον ιστότοπό μας επίσης. Και πέραν αυτού πιστεύω πως όλοι εμείς πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους γύρω μας για τα θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Και σίγουρα είναι μία από τις προτεραιότητές μου για το μέλλον. Και όσον αφορά τις γλώσσες, μεταφράζουμε σε όλες τις γλώσσες τις ετήσιες εκθέσεις μας. Υπάρχουν μεταφράσεις του παραρτήματος της ε, έκθεσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες, το οποίο δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα το έχουμε και πάλι στο μέλλον. Και πράγματι αυτό το λέω διότι με αφορά ιδιαίτερα, διότι η δική μου γλώσσα δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Και έχω πραγματικά επίγνωση του πόσο σημαντικό είναι να έχεις πληροφορία στη γλώσσα σου, γιατί η γλώσσα δεν είναι μόνο λέξεις, είναι και έκφραση του πολιτισμού σου. Γι' αυτό λοιπόν προστατεύοντας τη γλώσσα, προστατεύεις και τον πολιτισμό σου. Και όσον αφορά το φίλο, να σας πω ότι όταν έγινε διαμεσολαβήτρια στην Ιρλανδία ήταν η πρώτη ερώτηση που μου ετέθη. Ναι, διαμεσολαβήτρια και όχι διαμεσολαβητής. Και πάλι αυτό έχει σχέση με τον πολιτισμό. Ε, δεν θεωρώ τον εαυτό μου φεμινίστρια, Όμως όταν ερωτήθηκα για το θέμα αυτό στην Ιρλανδία, απάντησα ότι θα απαντώ και στην προσφώνηση κυρία Δημοσολαβήτη και κυρία Δημοσολαβήτρια. Βέβαια πολλά μέλη από τη Σουηδία εξέφερσαν τις αντιρρήσεις τους. Γι' αυτό ξέρω γιατί η λέξη διαμεσολαβητής είναι σουηδική ombudsman και αναφέρεται σε κάποιον άντρα. Και πραγματικά είναι εκπληκτικό όταν βλέπει κανείς πόσες διαφορές υπάρχουν στις κάθε γλώσσες. Κάποιες γλώσσες αναφέρονται σε διαμεσολαβητή, κάποιες γλώσσες σε υπέρμαχους των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Εγώ προσωπικά πάντα βλέπω τον διαμεσολαβητή όχι ως ε, υπερασπιστή ή συνήγορο οποιοδήποτε, αλλά ως όντως ένα, ένα μέσο διαμεσολάβησης ανάμεσα σε δύο άτομα. Εμείς προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε την, τις δυνάμεις ανάμεσα στο θεσμικό όργανο και στο άτομο και θέλουμε να κάνουμε το άτομο τόσο ισχυρό όσο και το θεσμικό όργανο και έχουμε στη διάθεσή του όλες τις δυνάμεις μας και όλες τις δυνατότητες για έρευνα έτσι ώστε το άτομο να μπορέσει να υποβάλει μια καταγγελία για αυτό που τον απασχολεί. Βέβαια φυσικά να τονίσω ότι δεν ασχολούμαστε με μια καταγγελία θεωρώντας ότι δίκιο έχει ο καταγγέλων. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω πως είμαστε αμερόληπτοι. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιλέξει να δώσει έναν ε, διαφορετικό ορισμό για το έργο μου, θα συμφωνήσω, δεν θα φτάσω μέχρι εκεί. Τώρα δίνω τον λόγο στην Μπέατρις Δεσέρα από την ομάδα Άλβερ. Νομίζω ότι είναι και η μοναδική λέξη την οποία γνωρίζω στη γλώσσα σας αυτό το οποίο είπατε πρόεδρε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την διαμεσολαβήτρια και θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους ότι το ότι είναι η μοναδική υποψηφία δείχνει πόσο σημαντική είναι η δουλειά σας μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια της μικρής περίοδου που είσαστε στη θέση αυτή, όπως είδαμε με την έκθεση που εγκρίναμε σήμερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι το, η υπηρεσία σας είναι μια ευρωπαϊκή υπηρεσία, είναι ένα ευρωπαϊκό όργανο και θα πρέπει ακριβώς να σεβόμαστε και να εξετάζουμε φυσικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε σαν μια συλλογική λειτουργία, σαν μια ομάδα η οποία ε, ε, πλαισιώνει κατά κάποιο τρόπο την δράση σας. Και μπορώ να πω ότι δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να ακούμε στα πλαίσια των κοινοτικών οργάνων, το ότι παλεύετε για την βέλτιστη δυνατή λειτουργία, για τη δημιουργία ομάδων οι οποίες είναι μονίμως στην υπηρεσία των, του κοινού και των πολιτών και την επιδίωξη γενικότερα της αριστείας των τρόπων λειτουργίας σας. Εδώ νομίζω ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι, κάτι, είναι κάποια που ενδιαφέρεται όχι μόνο στο να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά στο να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στην επικοινωνία, στους τρόπους επικοινωνίας που επιδιώκει ο πολίτης. Έχει σημασία λοιπόν να εργαστείτε ε, υπέρ της νομιμοποίησης του τρόπου με τον οποίο εργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με πλήρη διαφάνεια τα ευρωπαϊκά όργανα θα πρέπει να ενισχύσουν αυτήν την διαδικασία μονιμοποίησης απαραίτητης για τους πολίτες μας. Νομίζω ότι αυτό το είδος της ιδιότητας του υπαλλήλου την οποία έχουμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτούς οι οποίοι δεν είναι υπέρ του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούν, προβλέπεται να λειτουργούν οι υπηρεσίες μας. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως η σημερινή ε, στις χώρες μας οικονομικής αποσταθεροποίησης, διαφθοράς, μια πραγματικά δημοσιοϊπαλληλική αντίληψη σωστή και ε, αποτελεσματική είναι απαραίτητη για όλους. Έτσι θα διασφαλίσουμε λοιπόν ε, την ε, σωστή δεοντολογική λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. Τώρα, σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, θα ήθελα μόνο να θέσω μία ερώτηση προς την κυρία Ρέλη. Σε σχέση με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς στα πλαίσια της Επιτροπής Αναφορών αποφασίσαμε ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς, ο οποίος έχει μια τεράστια γάμα αρμοδιοτήτων, θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος θα αποτελεί, αν θέλετε, τον κατεξοχήν συνομιλητή μας, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και αυξάνοντας τις δυνατότητες επικοινωνίας. Δεν ξέρω πώς μπορούμε λοιπόν να συνδεθούμε και με την υπηρεσία του Ombudsman έτσι ώστε να λειτουργήσουμε με πιο σωστό τρόπο και θα ήθελα να μας πείτε εσείς τι ιδέες έχετε έτσι ώστε να συνεργαστείτε με την δημιουργία και με τον καθορισμό των όρων συνεργασίας με τον κύριο Τίμερμανς. Νομίζω προσωπικά λοιπόν είναι να μην ξεχάσουμε ε, να επικοινωνούμε αυτά τα οποία κάνουμε. Η ύπαρξη της υπηρεσίας σας είναι μεν σημαντική, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την επικοινωνία με στρατηγικό τρόπο. Τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να τα βελτιώνουμε, αλλά θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ε, στους πολίτες μας που είναι οι εργοδότες μας αν θέλετε, ε, πώς μπορούμε να τους μεταφέρουμε αυτά τα οποία κάνουμε. Ε, δεν ξέρω αν με το κοινωνικά δίκτυα, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έχει μεγάλη σημασία έτσι ώστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να επικοινωνήσουμε ε, και να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών. Όχι γιατί είμαστε πάρα πολύ σύγχρονοι, όχι γιατί είμαστε καλύτεροι από τους προκατόχους μας. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα, νέα και παλιά, έτσι ώστε να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή μας που είναι να προσδώσουμε νόημα και να καταστήσουμε αποτελεσματική τη διαδικασία κατάθεσης αναφορών από τους ε, συμπολίτες μας. Επιμένω λοιπόν τελειώνοντας ότι απαιτείται μια μόνιμη διασύνδεση ανάμεσα στη δική μας Επιτροπή και τη δική σας υπηρεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ε, χρήσιμα όλα αυτά για μένα. Ε, συμφωνώ μαζί σας ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ε, και όποτε μπορώ το ασχολούμαι με το θέμα αυτό και υπάρχουν ορισμένα σκάνδαλα τα οποία εμπλέκουν ορισμένους αξιωματούχους της Επιτροπής καμιά φορά και νομίζω ότι όλη η Επιτροπή και η Γραμματεία της Επιτροπής υποφέρει όταν υπάρχουν τέτοια σκάνδαλα. Εναπόκειται σε όλους μας να υποστηρίξουμε τους, τα στελέχη και να περάσουμε το μήνυμα, να πούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται έντιμα και αποδοτικά. Ε, συμφωνώ μαζί σας σχετικά με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς, είναι πάρα πολύ σημαντικός για αυτή την Επιτροπή και σημαντικός για το έργο του, της διαμεσολαβήτριας, ε, διότι το έργο του γίνεται σε ένα πλαίσιο πολιτικά ε, διότι είναι να υπάρχει ένα, μια ένας συνασπισμός ε, δυνάμεων που συνεργάζονται μαζί και οι προτάσεις που έγιναν πρόσφατα σχετικά με την ε, διαφάνεια ε, δεν ανεφίσανε επειδή κάποιος, εσείς, εγώ είπαμε κάτι, αλλά ήταν ένα σύνολο δυνάμεων που προσπαθεί να προωθήσει αυτό το θέμα. Το προσωπικό μου θα συναντήσει τον κύριο Τίμεμανς και μέλη του ε, γραφείου του και νομίζω ότι το βασικό μου μήνυμα προς αυτόν θα είναι ότι είμαστε και οι δύο ε, στο, στην ίδια, κάνουμε και δύο την ίδια δουλειά, αλλά η δική του δουλειά δεν είναι να υπερασπίζεται την Κομισιόν Πάση Θυσία και δική μου, το δικό μου έργο δεν είναι να κατακρίνει ε, σε κάθε περίπτωση την Κομισιόν. Πρέπει να μάθουμε να εργαζόμαστε με, συνεργα... με πνεύμα συνεργασίας ε, εκείνος και η Κομισιόν. Δεν λέω ότι δεν το κάνουν, αλλά πρέπει ίσως να βελτιώσουμε τους κανόνες συμμόρφωσης και να θεωρούν το γραφείο μου, την υπηρεσία μου ως κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει στην εργασία τους ε, και θα πρέπει να υποστηρίξουν τις αξίες που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν στα επόμενα πέντε χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό που σημαίνει αυτό είναι ότι ορισμένες τροχοπέδες που υπάρχουν ανάμεσα στο γραφείο μου και ε, στην Επιτροπή ορισμένα εμπόδια ε, όσον αφορά τις ε, περίεργες καταγγελίες που πρέπει να περνούν και πάρα πολλά από αυτά τα εμπόδια, τα μπλοκαρίσματα φαίνεται ότι είναι ένα είδος ένας φόβος μήπως αποκτήσουν κάποια εξουσία ορισμένα στελέχη χαμηλού επίπεδου ε, και μπορούν και έχουν επικοινωνία με το δικό μου ε, το γραφείο και την υπηρεσία. Πάρα πολύ συχνά δεν υπάρχει το είδος του διαλόγου που απαιτείται σε όλα τα επίπεδα ε, τις υπηρεσίες ούτως ώστε να περνούν αυτά τα μηνύματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσω μαζί του. Υπάρχει επίσης από το Κανάρι το, ε, σχετικά ε, με τα δηλητηριώδη αέρια που υπάρχουν στα ανθρακοριχεία. Κατά κάποιο τρόπο ο Ombudsman μπορεί να δράσει ε, για ούτως ώστε να μην πεθαίνουν άνθρωποι από δηλητηριώδη αέρια και θα πρέπει ε, να δούμε πού υπάρχει κακοδιοίκηση, κακοδιαχείριση ε, στις ε, υπηρεσίες της Κομισιόν. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική, μια άτυπη μορφή συνεργασίας όσον αφορά τις κατεγγελίες και τις έρευνες τις διοικητικές και τις προσφυγές μεγάλου δημοσίου ενδιαφέροντας. Νομίζω ότι θα μπορούμε μαζί να επιτύχουμε πολλά πράγματα. Ε, ελπίζω ότι θα αναπτύξω μεγάλη συνεργασία με τον Επίτροπο Τίμερμανς και με άλλους ε, επιτρόπους ε, και τις γραμματείες τους. Τη γραμματεία της Κομισιόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κόλσον. κυρία Κόλσον, όχι, δεν θέλει να λάβει τον λόγο. Σόλκον, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Έμιλι, για την καλή δουλειά σου μέχρι τώρα. Αν ε, αισθάνεσαι όπως αισθανόμαστε πέρσι ε, το θέρος, ότι είμαστε ασφαλείς που μπορούμε να σε συστήσουμε ε, στο Κοινοβούλιο. Και θα μπορούσα να πω εδώ να τονίσω ότι η διαφάνεια και η συμμετοχή των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα εστιαστώ λίγο σε ένα θέμα. Πάρα πολλές φορές έχω αναφερθεί σε υποσχέσεις που υπάρχουν στη συνθήκη ότι θα έχουμε μια καλή διοίκηση ασφαλή ε, και συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Με καλή διοίκηση εμείς ε, του, τουλάχιστον που είμαστε από τον Βορρά ε, σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι μια βασική αρχή της υπηρεσίας που προστατεύει τους πολίτες, όχι μόνο τους ε, δημόσιους υπαλλήλους. Βεβαίως και προστασία των δημοσίων υπαλλήλων που θα πρέπει να έχουν περισσότερη αξιοπρίπεια στην ε, δουλειά τους ε, παρά όταν καλύπτονται από την δίκηση. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και είναι καλύτερα μέσα καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτό πώς θα μπορούσαμε να βεβαιωθούμε με την πρόταση αυτή θα έχουμε έναν κανονισμό για καλή διαφάνεια, διότι υπάρχει το θέμα εδώ και, εδώ και καιρό. Έχετε κάποια εντύπωση ότι θα γίνει κάτι. Εγώ θα προτιμούσα να μην έχουμε κατευθυντήριες γραμμές, αλλά να έχουμε έναν κανονισμό. Δεύτερον, πώς νομίζετε ότι όλο ε, το, θέμα ε, του συμφέροντος ε, καλύπτεται διότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για τα θεσμικά όργανα να αντιληφθούν ότι η σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα κριτήριο αντικειμενικό. Δεν μπορείτε να απαλλαγείτε μετά από τα συμφέροντά σας απλώς δηλώνοντάς σας και να πούμε για κάποιον ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, θα πρέπει να είναι αντικειμενικό, να, υπάρχει, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για σύγκρουση συμφερόντων όταν ε, λαμβάνονται αποφάσεις εκ μέρους των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό έχει αναγνωριστεί από τα θεσμικά όργανα και έχω την εντύπωση ότι η ΕΦΣΑ, η ΕΜΑ, οι διάφορες οργανισμοί το έχουν καταλάβει αυτό. Αυτή είναι η περίπτωση στη Δανία και σε πάρα πολλές χώρες. Νομίζουν όμως αλλού πολλοί ότι αν δηλώσει κανείς τα συμφέροντά του αυτό αρκεί και ότι δεν υπάρχει σύγκρουση. Όχι, όχι, δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος αυτός και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς το όλο θέμα. Και το τρίτο σημείο, κατά τη γνώμη μου, λιγότερο ενδιαφέρον, αλλά ε, παρόλα αυτά πώς εμείς στο Κοινοβούλιο μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας δίνοντας πρόσβαση στους πολίτες. Είμαστε αρκετά διαφανείς εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο. Σοκαρίστηκα όταν ο πρόεδρος αποφάσισε ότι ε, υπογραφή για σύσταση, για όμπουτσμαν πρέπει να παραμείνει μυστική. Έχουμε μυστικές ψηφοφορίες, αλλά εμείς ε, βάζουμε όλο το κύρος μας πίσω από κάποια σύσταση ως ευρωβουλευτές. Γιατί λοιπόν για τους πολίτες ε, να είναι μυστικές αυτές οι υπογραφές, απόρριτες. Και γενικά πιστεύετε ότι βεβαίως έχουμε διαφορετικά καθήκοντα από ό,τι τα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά παρόλα αυτά και από ό,τι σας θυμάμαι είσαστε η μόνη ombudsman που έχετε το δικαίωμα να κατακρίνετε και το κοινοβούλιο να επικρίνετε το κοινοβούλιο σε άλλες χώρες. Το κοινοβούλιο βρίσκεται πιο πάνω και δεν μπορεί να επικρίνεται από τον ε, διαμεσολαβητή. Αν έχετε το δικαίωμα, έχετε και το καθήκον να μας κρίνετε εάν δεν κάνουμε αυτό ε, που πρέπει να κάνουμε αν δεν μεταχειριζόμαστε τους πολίτες ε, με τον τρόπο που πρέπει, αν δεν τους εμπλέκουμε ε, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ε, βεβαίως, το θέμα των υπογραφών επίσης είναι σημαντικό, αλλά βεβαίως δεν πρέπει εμείς να καλυπτόμεθα και να κρυβόμαστε από την γνώση των πολιτών, ορθώνοντας περίεργους τείχους και τείχη για να κρύψουμε τα λάθη μας, να καρτούμε μυστικά από τους πολίτες. Και νομίζετε ότι εμείς είμαστε στο ύψος των δικών σας προσδοκιών. Είμαστε ο κατάλληλος εταίρος για την συμμετοχή των πολιτών και τη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Άουκεν για τα καλά σας λόγια στην αρχή και για τις ερωτήσεις σας. Πράγματι, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολλές εκθέσεις και πολλές θέσει για μια πιθανή νομοθεσία περί ευρωπαϊκής διοίκησης. Δεν προχώρησε πολύ το θέμα αυτό και πιστεύω ότι τελευταία, το τελευταίο κοινοβούλιο δεν είχε αρκετή πολιτική θέληση έτσι ώστε να πιέσει για να, για να δρομολογηθεί το θέμα. Και εμείς προσπαθήσαμε σε πιο ακαδημαϊκό επίπεδο και υπήρχαν κάποιες επαφές ανάμεσα στο δικό μου γραφείο και σε μια ομάδα πανεπιστημιακών έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντάξουμε έναν κώδικα διατολογία για την Ευρωπαϊκή Διοίκηση. Και υποθέτω πως πάλι, όπως και πριν, εξαρτώμαστε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τους αρμόδιους επιτρόπους για να δρομολογηθεί το θέμα αυτό. Διότι καταρχάς όλοι ξέρουμε πού θέλουμε να βρισκόμαστε σε, στην ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά το πώς θέλουμε να διοικούνται τα θεσμικά όργανα και αυτή την περίοδο υπάρχει έτσι μια μεγάλη ποικιλία πρακτικών και προτύπων στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση. Του χρόνου κλείνουν 20 χρόνια από τη δημιουργία της θέσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και θα διοργανώσουμε ορισμένες εκδηλώσεις. Θα έχουμε μία εκδήλωση όπου θα δούμε αναδρομικά τα 20 χρόνια λειτουργίας του θεσμού αυτού και μετά θα συζητηθούν ακριβώς αυτά που αναφέρατε. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν εμείς αρχικά να κάνουμε την αυτοκριτική μας προτού προχωρήσουμε στα άλλα θεσμικά όργανα και φυσικά πρέπει όλοι να συμμετέχουν και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Τώρα όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνες σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιπτώσεις συγκρούσης συμφερόντων όταν ανώτεροι αξιωματούχοι καταλείπουν την, ε, το ευρωπαϊκό δημόσιο και πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε 55 φακέλους τέτοιων περιπτώσεων και κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή πώς αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις περιπτώσεις αυτές και αν επαρκεί ο κώδικας διοντολογίας έτσι ώστε να εντοπιστεί μία ανάρμοστη συμπεριφορά και να επιβληθούν κυρώσεις. Έχουμε κάνει συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το πώς να βελτιωθεί η συμμόρφωση και ανάμεσα σε αυτές τις συστάσεις ήταν για παράδειγμα ότι όσοι κάνουν αίτηση, όσοι ανώτεροι αξιωματούχοι κάνουν αίτηση να μεταβούν στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να είναι ανεξά, θα πρέπει η θέση που θέλουν να, ε, στην οποία θέλουν να πάνε να μην έχει καμία σχέση με την αρμοδιότητα που είχαν στην, στο ευρωπαϊκό δημόσιο. Και μια άλλη σύσταση που είναι έτσι ίσως προκλητική είναι όταν ανώτεροι αξιωματούχοι μεταβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα τα ονόματά τους να καταγράφονται σε ένα δημόσιο μητρό. Δηλαδή, αν εγώ, για παράδειγμα, η Emily O'Reilly θέλω να φύγω από αυτή τη θέση και να πάω να δουλέψω στην Coca-Cola, παράδειγμα, δεν ισχύει, αυτό να καταγράφεται, να αναγράφεται δηλαδή τι ακριβώς δουλειά έκανα στην ε, γενική διεύθυνση στην οποία βρισκόμουν και τι δουλειά προτίθαμε να κάνω στην ιδιωτική επιχείρηση. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την... Και επίσης το σκεπτικό πίσω από αυτήν την απόφαση που έλαβα και οι περιορισμοί που θα πρέπει να έχω. Φυσικά αυτό προσδίδει μεγαλύτερη διαφάνεια και αναγκάζει τους ε, ανώτερους αυτούς αξιωματούχους που θέλουν να αποχωρήσουν να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές. Αυτό πιστεύω πως είναι και προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι αργά ή γρήγορα οι πολίτες θα ανακαλύψουν τι συμβαίνει. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, τη European Voice, έχουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τη Transparency International ας πούμε. Γίνεται λοιπόν, μαθεύονται αυτά τα πράγματα, όμως θα ήταν πιο απλή και γρήγορη διαδικασία εάν από τα ίδια τα θεσμικά όργανα υπήρχε μια, ένα τέτοιο μητρό, ένα τέτοιο κατάλογος έτσι ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Πιστεύω πως ε, όλοι μας συμμεριζόμαστε την ίδια άποψη για τη σύγκρουση συμφερόντων, αλλά όπως είπα και στην αρχή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να θέσουν ψηλά τον πύχη και να έχουν τα υψηλότερα και αυστηρότερα δυνατά πρότυπα. Και να επαναλάβω σε αυτό το σημείο ότι ανυπομονώ να, αρχίσω να συνεχίσω μάλλον τη συνεργασία μου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Και σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά και μπορώ να σχολιάσω, να τοποθετηθώ και να κάνω σχόλια για τη διοίκηση του Κοινοβουλίου και θα το κάνω όπως το έκανε και ο προκάτοχός μου. Θα σας ασκήσω λοιπόν κριτική. Πιστεύω όμως πως ε, το έργο σας είναι κάτι διαφορετικό και πιστεύω πως εσείς έτσι κι αλλιώς έχετε έναν κώδικα δεοντολογίας ο οποίος υποθέτω πως έχει συνταχθεί από τη γραμματεία μετά από διαβουλεύσεις και πρόσφατα Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση του Κλάους Βέλε, του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναφέρει τρόπους με τους οποίους θα γίνει πιο αποτελεσματικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω πως εκεί υπάρχουν ορισμένες και σωστές προτάσεις όσον αφορά τη διαφάνεια και την αντιμετώπιση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Βέβαια είμαι σίγουρη πως θα το παρακολουθείτε και εσείς ε, στενά. Θέλω να πω όμως ότι όταν εσείς λαμβάνετε καταγγελίες οι οποίες εμπίπτουν στη δική μου αρμοδιότητα και δεν είναι πολιτικού χαρακτήρα, ναι, φυσικά θα ασχοληθώ με αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μακάρθη από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα. Δεν είμαι μέλος τακτικό της Επιτροπής σας, θα ήθελα όμως να είμαι εδώ σαν Ιρλανδός βουλευτής και καταρχάς να συγχαρώ την Έμιλι Ράιλι για την εξαιρετική δουλειά την οποία είχε επιτελέσει από τότε που ανέλαβε η υπηρεσία και να ευχηθώ να εξελιχθεί σωστά η διαδικασία εκλογής της. Από ό,τι φαίνεται τα καταφέρνει η Έμελη και φόβησε όλους τους αντιπάλους της, τους ανταγωνιστές της και έμεινε μόνη της υποψηφία. Μία ερώτηση σχετικά με το TTIP και τη διαβούλευση για το TTIP. Αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία είπατε είναι ότι ήδη υπάρχουν ε, πάρα πολλές αναφορές γύρω από το θέμα αυτό και δεν το είχα υπόψη μου. έχει πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να γίνει πιο ανοιχτή, έχει αποφασίσει η, Ευρω... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει πιο α, διαφανής και ειδικότερα για το TTIP και γενικότερα. Νομίζω ότι υπήρξε μια προσπάθεια να είναι πιο ειλικρινής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα που εμπλέκονται στις διαδικασίες του TTIP. Πρέπει να είναι πιο δεκτική και πιο διαφανής. Υπάρχει επίσης και μία πρωτοβουλία των πολιτών, η οποία φτάνει περίπου το 1 εκατομμύριο σε σχέση με τον μηχανισμό EISTS. Ε και η οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην συμπεριληφθούν ορισμένα πράγματα στις συνομιλίες. Λοιπόν, τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε να εξετάσετε αν έχουν συλλεγεί επαρκή αριθμοί υπογραφών και σε ποιο βαθμό μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγνοήσει αυτές τις ε, προσπάθειες συλλογή υπογραφών. ιδιαίτερα σε χώρες όπου υπάρχει επιφυλακτικότητα σαν τη δική μας που χρειάστηκε να ψηφίσουμε τη συνθήκη δύο φορές. Λοιπόν, δεν είναι τόσο γραφειοκρατική η υπηρεσία μου, αν θέλεις να συνεισφέρεις, ε, σου. Τώρα για το TTIP. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι θέλει να είναι πιο δεκτική, πιο διαφανής. Έχουμε κάνει ε, πρόσθετες επιπλέον προτάσεις και σε σχέση με το ISDS το θέμα είναι πολιτικό, θα εξαρτηθεί από πάρα πολλούς. Έχουν οργανωθεί κάποιες ακροάσεις, έχω έρθει σε επαφή και με την κυρία Μάλστρομ. Ο ρόλος μου δεν είναι να λέω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα δέχεστε αυτό ή εκείνο ρόλος μου είναι να ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ασχολείται με κάποια θέματα να το κάνει αποτελεσματικά αλλά και με διαφάνεια και κρατώντας πάντα τα συμφέροντα του Ευρωπαίου πολίτη ε, στο κέντρο των ενδιαφερόντων της. Τώρα, αν ένα εκατομμύριο πολίτες υπογράφουν ε, μια αναφορά, προφανώς αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά ε, υπόψη. Δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ συνοπτικό τρόπο και αυτοί που υπέγραψαν τη συγκεκριμένη αναφορά πρέπει να αναγνωρίσουν τη μεγάλη προσοχή η οποία δόθηκε στο αίτημά τους. επικοινωνία ανάμεσα σε αυτούς τις ομάδες που έχουν υπογράψει με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο κτλ. έτσι ώστε όλες οι εξηγήσει που δίδονται να είναι σωστά τεκμηριωμένες και να έχει προηγηθεί επαρκές ποσοστό διαβούλευσης. Δεν έχει φτάσει ακόμα το 1 εκατομμύριο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το πολιτικό καθαρά. Το θέμα είναι να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα με σοβαρό τρόπο και να μην αγνοήσει το τι επιζητεί στην παρούσα φάση ένα εκατομμύριο κόσμος. Τώρα σε σχέση πάντα με το TTIP και την διαπραγματευτική εντολή. Θα δείτε ότι είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί ακόμα και στην ιστοσελίδα μου. Θα δείτε ότι είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πάντως θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να μην είναι πολύ επιφυλακτικά θα πρέπει να αρχίσουν να εμπιστεύονται τους πολίτες περισσότερο από ό,τι σήμερα. Μερικές φορές τα θεσμικά όργανα ε, προσπαθούν να παίρνουν αποφάσεις ξεκάθαρες, ε, κάνουν, δεν κάνουν διακρίσεις, δεν κάνουν θα έλεγα τις απαιτούμενες, δεν μπαίνουν στο απαιτούμενο, ε, στις απαιτούμενες λεπτομέρειες για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν. Λοιπόν, θα πρέπει να διευκρινίσουμε στους πολίτες τι ακριβώς μπορεί να συμβεί στην περίπτωση ε, κατά την οποία ε, δημοσιοποιηθεί μια, ε, ένα κομμάτι των διαπραγματεύσεων και ακόμα και αν υπάρξει κάποια συσσαγωγικά βλάβη γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουν να το αντισταθμίσουν κατά τη διάρκεια πάντα των ίδιων διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να κάνουν περισσότερα πόσο όσο έχουν κάνει. Έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σε επίπεδο διαφάνειας και θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες. Σίγουρα πάντως έχουν κάνει βήματα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι το τέλος του καταλόγου των ομιλητών. Εγώ είμαι τελευταία, είμαι ίσως σε μειονεκτική θέση, διότι πάρα πολλές από τις ερωτήσεις έχουν τεθεί. Ευχαριστώ πολύ και για τις απαντήσεις. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, έχετε το λόγο. Ευσάκη πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντήσαμε και πάλι, κυρία Διαμεσολαβήτρια και με την ευκαιρία της ακροασής σας για μια νέα θητεία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δουλειά σας και την δέσμευσή σας να ενισχύσετε τα δικαιώματα των πολιτών. Ε, διάβασα το έγγραφο για τη νέα ε, στρατηγική και με βάση το έγγραφο αυτό έχω δύο σύντομες ερωτήσεις να σας απευθύνω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσος διαμεσολαβήτρια βλέπετε το μέλλον ε, της ε, πρωτοβουλίας των ε, πολιτών γενικά. Το 2015 θα είναι η αναθεώρηση του κανονισμού για την πρωτοβουλία και το Κοινοβούλιο ετοιμάζει έκθεση και ακρόαση για το θέμα και εσείς κάνετε έρευνα σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή και τα συμπεράσματά σας θα μας βοηθήσουν για την δική μας έκθεση. Και δεύτερον, ξέρω ότι δεν είναι ρόλος ε, της διαμεσολαβήτριας ε, σχετικά ε, με την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σας πώς αυτό θα αλλάξει τον τομέα δραστηριοτήτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις δύο ερωτήσεις σε σχέση με την πρωτοβουλία των πολιτών Έχουμε αρχίσει μια εξέταση, μια έρευνα και ο κύριος, τα σχόλια του κυρίου Τίμερμανς είναι σημαντικά. Υπάρχει κίνδυνος εάν έχουμε διαφορετική προσέγγιση, ε, πιο ε, πολιτική ή λιγότερο νομικίστικη, υπάρχει κίνδυνος και στις συναντήσεις με αξιωματούχους της Κομισιό ε, τους ενθαρρύνουμε, όπως είπα, να μας διαβουλευθούν ε, όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Η περίοδος ε, είναι πολύ σύντομη, τρεις μήνες και υπάρχει ε, ανάγκη αλλαγής ίσως στον κανονισμό. Και απαντώντας σε μένα που διάβασα εν συντομία ότι χαιρετίζουν τη δική μου σύσταση και πρόταση ως μέρος της δικής τους αναθεώρησης και ελπίζω ότι θα, όταν έχω τον Ιανουάριο ε, αυτά τα συμπεράσματα θα μπορέσω να συμβάλλω στη δική σας δουλειά. Σε σχέση με τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ξέρω τη συζήτηση που λαμβάνει η χώρα. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και έχω κάνει και έρευνα σχετικά με το πώς οι πόροι του Ταμείου Συνοχής ξοδεύονται στα κράτη-μέλη. Οι διαδικασίες της Κομισιόν ούτως ώστε αν τα, οι δαπάνες αυτές είναι σύμφωνες, συμβατές με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Βεβαίως θα πρέπει να ενσωματώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις πολιτικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ε, καλό και θα πρέπει να δούμε τα, ποια είναι τα αποτελέσματα πολλών από αυτές τις συμβάσεις. Αυτό που προσπαθώ να κάνω στη δική μου δουλειά είναι να συνδέσω με πρακτικό τρόπο τα διάφορα άρθρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα άτομα με αναπηρίες για να δούμε ε, πώς εφαρμόζονται στα θεσμικά όργανα και μόνο με αυτήν την πρακτική εργασία θα δούμε ποια είναι η πραγματική αξία του χάρτη και των εγγράφων αυτών. Έχουμε ένα, ε, ένα νέο αίτημα για... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Έχω μία ερώτηση και μία, μία, μία πρόταση. Διαπίστωση. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί και ότι υπάρχει μία υποψήφια αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολες οι αρμοδιότητες ε, του διαμεσολαβητή και γι' αυτό υπάρχει ένας υποψήφιος ή ότι εργαστήκατε πάρα πολύ καλά και αυτό είναι ο λόγος που σας εμπιστευόμαστε εκ των προτέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξάλλου εξεπλάγει που ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου αποφάσισε ότι οι υπογραφές μας δεν θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν αν σας υποστηρίξουμε αυτό. Είναι παιδιάστικο αν υπογράφω κάτι θα πρέπει ε, να γίνεται για να δημοσιοποιείται. Δεύτερον, ε, η πρόταση εργαζόμαστε από την ίδια πλευρά για τους πολίτες και τα δικαιώματά τους και η Επιτροπή Αναφορών το τελευταίο καιρό έχει ένα πρόβλημα θα έλεγα είναι ε, δύσκολο να περάσουν τα δικαιώματα της πρόκειται για τα παιδιά. Τα παιδιά δυσκολεύονται να στραφούν ή να καταφύγουν, να προσφύγουν ε, σε ένα θεσμικό όργανο. Είναι μια ιδέα για τις μελλοντικέ εργασίες, διότι στην τελευταία συνάντηση είχαμε φακέλους όπου είχαμε ένα μπλοκάρισμα. Ίσως είναι μια γραμμή που θα μπορούμε να δούμε μαζί και να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρχει μια καλύτερο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάρ για τα καλά σας ε, σχόλια. Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ σε αυτήν εδώ την Επιτροπή καλεσμένους ε, διαμεσολαβητές για τα παιδιά. Πιστεύω πως είναι ένα πολύτιμο έργο που κάνουν και Πώ έχουν να μας διδάξουν πολλά. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, πράγματι θα ήταν καλή ιδέα να τους ε, καλέσετε. Έχω συζητήσει με συναδέλφους και ξέρω πόσο δύσκολα είναι αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κρατήσει την τελευταία θέση για μένα. Τώρα θα κάνω την ερώτησή μου και μπορείτε να ολοκληρώσετε. Όπως είπα, σας έγιναν πολλές ερωτήσεις και τις απαντήσατε. Καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ διότι όσον καιρό ήσασταν στη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχετε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και πιστεύω πως είμαστε όλοι ικανοποιημένοι από το έργο σας και είμαστε σίγουροι ότι θα έχετε πάρα πολύ χρόνο για να συνεχίσετε αυτά που έχετε αρχίσει και να τηρήσετε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχετε δώσει. Μετά από όλα όσα είπατε για τη διαφάνεια, για την ορατότητα και για την επικοινωνία, πρέπει να πω ότι αυτό που επιθυμεί ο πολίτης είναι να αισθάνεται ότι είναι κοντά στα θεσμικά όργανα και ότι γίνεται ακουστός. Και αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων και μέσω μιας ε, γρήγορης απάντησης δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι από τον χρόνο απάντησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν έχετε σκοπό να μειώσετε τη γραφειοκρατία όπως έχετε πει και το πώς σκοπεύετε να το κάνετε αυτό έτσι ώστε να γίνετε πιο αποτελεσματικοί και πώς θα το δείξετε αυτό στους πολίτες. Και μετά μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Πράγματι, έχετε δίκιο. Θα έχετε τη δυνατότητα να με ελέγχετε για αρκετό καιρό. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τα σχόλια και σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα το μέλλον. Βέβαια μου αρέσει αυτό και φυσικά και δέχομαι να υποβληθώ και εγώ σε έλεγχο όπως και εγώ υποβάλλω τα θεσμικά όργανα σε έλεγχο είναι μέλο, μέρος των αρμοδιοτήτων μου και πιστεύω πως αυτό με βοηθά έτσι και αλλιώ στο να βελτιωθώ και να βελτιώσω και την ποιότητα του έργου μου. Το ζήτημα που αναφέρεται είναι κάτι που απασχολεί το γραφείο του Διαμεσολαβητή εδώ και καιρό και πιστεύω πως και την, και την Επιτροπή Αναφορών αλλά και άλλες επιτροπές όντως πρέπει να επιταχύνουμε το έργο μας και το χρόνο απάντησης. Η εμπειρία μου εδώ τον τελευταίο χρόνο και τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ιρλανδία έχει δείξει ότι πραγματικά η αρχή της διαδικασίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν δηλαδή δεχόμαστε, λαμβάνουμε μια καταγγελία. Πρέπει ο τρόπος να είναι σωστός, διότι αυτό βοηθά και την υπόλοιπη διαδικασία. Την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα κατά το οποίο δεν αποφασίζει κανείς ad hoc για την μεταχείριση μιας καταγγελίας, μιας υπόθεσης, αλλά όπου υπάρχουν τρία διαφορετικά μέρη τα οποία θα συνδιαλλαγούν για το τι κατάληξη θα έχει μια καταγγελία και αφού εξεταστεί κάθε υπόθεση με λεπτομέρεια θα αποφασιστεί ποια πορεία θα ακολουθηθεί. Σίγουρα είναι προς το συμφέρον όλων μας μία πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική διαδικασία, αλλά όπως είπα και πριν είναι πολύ σημαντικό η επίσπευση αυτή της διαδικασίας να λάβει χώρα στην αρχή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα ολοκληρώνοντας να πω ότι ήταν μεγάλη μου χαρά που μπόρεσα να βρεθώ ενώπιόν σας. Μάργαρετ μη θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη προσοχή που δείχνετε όχι μόνο σε εμένα αλλά και στον ίδιο τον ε, θεσμό διότι χωρίς εσάς, χωρίς αυτήν την Επιτροπή να μας δίνει δύναμη δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το έργο μας με τον ίδιο τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για όλα όσα έχετε κάνει. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ήταν χαρά μας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή Αναφορών θα λάβει χώρα τέλη Ιανουαρίου, 25-26 Ιανουαρίου του 2015.